Αγαπητοί συνάδελφοι, προτείνω να αρχίσουμε αυτήν την τελευταία συνεδρία της Επιτροπής μας πριν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Είμαστε στο σημείο 12 της ημερήσιας διάταξης. για να ακούσουμε την παρουσίαση της μελέτης εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής, πρόθεση των εργασιακών και κοινωνικών προτύπων και η Ευρωπαϊκή Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. Δεν είναι φοβερό στα γαλλικά ο τίτλος. Λοιπόν, θα έλεγα καλύτερα κοινωνική ευθύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Ο κύριος Βέρνερ Άισχορτ ε, από την ε, Ίζα ε, και η κυρία Ντόριτ Βαλμπρίνκ από την Ήρας ενός Γερμανικού Ινστιτούτου Εργασίας και η Ίζα είναι ένα δανέζικο ιστιτούτο Ανάλυσης και Στρατηγικής. Αυτό, αυτή η μελέτη εκπονήθηκε στα πλαίσια μίας μελέτης που ο Ρίτσαρντ ζήτησε θα είστε εσείς ο πρώτος ομιλητής βεβαίως Αξιότιμοι βουλευτές, αγαπητοί πρόεδρε, θα Ήθελα να σας παρουσιάσω μια εξαιρετικά διεξοδική μελέτη για την εξωτερική διάσταση της, Ευρωπαϊκής, της κοινωνικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα σας ε, μοιράσω, θα μοιράσουμε την παρουσίαση ανάμεσα στους συναδέλφους. Ο συνάδελφός μου, ο κ. Βέρνερ Χάιχολς, θα σας κάνει την αρχική ε, παρουσίαση του ζητήματος. Στη συνέχεια θα μας μιλήσει για την συνοχή της εξωτερικής διάστασης κοινωνικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης η κυρία Ντορίτ Βαλμπρίνκ. Ε, και θα σας μιλήσει και για την αξιολόγηση αντικτύπου σχετικά με τα εργαλεία και τα μέτρα που χρησιμοποιήσαμε για να αξιολογήσουμε την κατάσταση σε διάφορες χώρες και μετά θα επανέλθω κι εγώ για κάποια ζητήματα πολιτικής. Ο Μάικλ Κέντζια θα σας κάνει την ε, παρουσίαση του ζητήματος, ε, θα παρουσιάσει το πρώτο τμήμα. Ε, πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο κεφάλαιο της παρουσίασής μας ε, θα ήθελα να σκιαγραφίσω το βασικό χαρακτήρα της εξωτερικής διάστασης της κοινωνικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναλύει η μελέτη την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρατηρεί ποιε ήταν οι τελευταίες εξελίξεις και αξιολογεί τον αντίκτυπο ε, της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκή Ένωση επί των τρίτων χωρών, των κρατών μη μελών της Ευρωπαϊκής ε, ο στόχος είναι να προωθηθούν πρότυπα εργασίας σε χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, οι συνθήκες εργασίας και τα εργατικά δικαιώματα είναι τα βασικά εστιακά σημεία της εσωτερικής και εξωτερικής κοινωνικής πολιτικής. Μέσα σε αυτή τη μελέτη καλύπτουμε ε, διάφορα θέματα προτεραιότητες για την περίοδο 2009-2010. Από τις αρχές του 1990 ε, έγιναν διάφορες πρωτοβουλίες ούτως ώστε να ενσωματωθούν σε εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποιες βασικές πολιτικές της Ένωσης στον τομέα αυτό. Στο σχεδίο δράσης από το 1995 έως το 1997 Ευρωπαϊκή Επιτροπή τόνισε ότι υπάρχει μία ανάγκη να τονίσουμε ε, και να δώσουμε έμφαση στην εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το κοινωνικό πρόγραμμα δράσης από το 2000 από το 1998 μέχρι το 2000 ε, εστίασε στις ε, βασικές ε, πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίστηκε η αυξανόμενη σημασία της εξωτερικής διάστασης Στη συνέχεια, το 2000, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατύπωσε την, ε, το κοινωνικό θεματολόγιο, το θεματολόγιο της κοινωνικής πολιτικής ε, και ασχολήθηκε με την εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Εστιάσαμε ε, στην ανταγωνιστικότητα, στην καινοτομία, στην αυξημένη κοινωνική συνοχή. Ήταν εξαιρετικά φιλόδοξη η πολιτική και το θεματολόγιο που εκπώνησε τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορεί να θεωρηθεί ως μια πειρά να δοθεί σφαιρική απάντηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκοσμιοποίηση και ε, τονίζεται έτσι η στενή σχέση ανάμεσα στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο και σε ιστορικό και σε εξωτερικό επίπεδο. Υπό το φως της αυξανόμενης παγκοσμιοποίησης ε, και αλληλεπίδρασης και αλληλεσύνδεσης όλων των κρατών, ε, προέκυψε σαφώ η ανάγκη να ενισχύσουμε την εξωτερική διάσταση τη κοινωνική πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, για να ε, ε, συνεισφέρουμε κι εμεί στον προγραμματισμό για την αντιμετώπιση τη παγκοσμιοποίηση χρησιμοποιώντα τα βιώματα και τι εμπειρίε Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να σα μιλήσω για την εσωτερική και εξωτερική διάσταση θα χρησιμοποιήσω μία παρομοίωση. Με τον πυρετό του παγκοσμίου κυπέλου η εσωτερική διάσταση θα μπορούσε να θεωρηθεί ω ένα αγώνα ε, στο γήπεδό μας ε, και αντίστοιχα η εξωτερική διάσταση ε, εκτός γήπεδου. Οπότε δεν είναι με εσά το κοινό αν θέλετε, δεν υποστηρίζεται η ομάδα σας όταν μιλάμε για την εξωτερική διάσταση. Το 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποίησε αυτή την κοινωνική ατζέντα το 2005 και την ανανεωμένη κοινωνική ατζέντα του 2008 για να εκπονήσει τη νέα πολιτική της. Να αναφερθώ εδώ στις πρόσφατες εργασίες της Επιτροπής με την έκθεση που εκπώνησε για την κοινωνική εταιρική ευθύνη στις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες. Στο δεύτερο τμήμα της παρουσίασης ε, θα θέλαμε να εστιάσετε την προσοχή σας στις κοινέ πρωτοβουλίες σχετικά με την εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, όπως προανέφερα, ε, ο, ο πυρήνα τη εξωτερική διάσταση κοινωνική πολιτική είναι οι δράσει ε, για την προώθηση τη αξιοπρεπού εργασία ε, και των εργατικών προτύπων σε χώρε που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βασικά πρότυπα, αξιοπρεπεί συνθήκε εργασία, προγράμματα αναχώρα, κοινωνική εταιρική ευθύνη, όλα αυτά είναι αναπόσπαστα και βασικά στοιχεία, συστατικά στοιχεία τη εξωτερική διάσταση. Στη διαφάνεια 10 τώρα βλέπουμε την ε, κοινωνική στρατηγική για την εξωτερική διάσταση που στην αρχή επικεντρώθηκε στη συζήτηση περί της κοινωνικής ρήτρας, δηλαδή να υπάρχουν κοινωνικές προϋποθέσεις ε, στις εξωτερικές σχέσεις και να ανταμείβονται οι χώρες που τηρούν ε, τα πρότυπα, χορηγώντας τους πλέον ευνοϊκές εμπορικές συμφωνίες. Από το 2001 και μετά η Ευρωπαϊκή Ένωση άρχισε να χρησιμοποιεί και άλλου είδους εργαλεία και μηχανισμούς για να προωθήσει τα κοινωνικά πρότυπα σε χώρε μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο στόχο είναι πάλι τα βασικά ε, εργατικά πρότυπα, αλλά έχουν ε, ε, ανανεωθεί τα εργαλεία, χρησιμοποιεί το διάλογο, χρησιμοποιούνται οι διαπραγματεύσει στο διεθνέ Γραφείο εργασία, παραδείγματο χάρη θεωρήθηκε ότι ήταν καλύτερος τρόπος αυτός για να προαγάγουμε ε, τα πρότυπα εργασίας. Στη διαφάνεια 11 έχουμε τον πίνακα με όλα τα εργαλεία που χρησιμοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να τα ταξινομήσουμε ως ε, σκληρά, μάλακα και ε, ε, χρηματοοικονομικού χαρακτήρα εργαλεία στις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, θα ασχοληθώ με τις εξωτερικές πολιτικές, δηλαδή με τη δεξιά ε, κολόνα, τη δεξιά στήλη. Είναι οι συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου, οι προτιμησιακές συμφωνίες GSP και GSP SIN και επίσης η προσέγγιση του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου ανήκει στα σκληρά εργαλεία. Επίσης ο διάλογος βλέπετε στο δεύτερο τετραγωνίδιο, τα κίνητρα, οι συστάσεις συνιστούν ε, μαλακά εργαλεία, ήπια εργαλεία. Ε, κατόπιν ε, βλέπετε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια και η τεχνική αρρωγή ταξινομούνται στα, μεταξύ των οικονομικών εργαλείων. Η συνοχή τώρα της εξωτερικής διάστασης. Όλο ένα και περισσότερο η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί τα ήπια εργαλεία και τώρα ολοκληρώνοντας ε, την δική μου παρουσίαση θα δώσω το λόγο στη συνάδελφο από τη Δανή για να παρουσιάσει το δικό της ε, κομμάτι. Εκτός Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Θα σας αναφέρω πρώτα την ανάλυση της ε, συνοχής της εξωτερικής διάστασης και κατόπιν θα σας μιλήσω για τα μέσα που έχουμε χρησιμοποιήσει. Όσον αφορά την ε, συνοχή έχουμε αναφέρει τρεις διαφορετικές ε, διαστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια τέτοια πολιτική. Η πρώτη διάσταση είναι η οριζόντια συνοχή όταν εξετάζουμε διάφορους τομείς πολιτικής. Έχουμε την κοινωνική πολιτική, την πολιτική εμπορίου και την αναπτυξιακή βοήθεια. Έχουμε δει λοιπόν αυξανόμενο βαθμό συνοχής. Το εμπόριο όμως είναι ο βασικός στόχος εδώ πέρα και αυτό επηρεάζει την εξωτερική διάσταση και την εξωτερική πολιτική. εξετάζοντας την κάθετη συνοχή, το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση προσεγγίζει διεθνείς ε, φορείς και πώς τους επηρεάζει. Δύο οργανώσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές, ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και ο ΠΟΕ. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρή επιρροή εντός του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, του ILO, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, ενεργεί πάντα ως ενιαίος φορέας και αυτό μερικές φορές δημιουργεί προβλήματα. Είναι όμως ε, σημαντικό φόρμα για τη συζήτηση των θεμάτων αυτών ε, το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Ο ΠΟΕ, στον ΠΟΕ είναι σαφές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας ενιαίος φορέας, ωστόσο δεν πρόκειται για φόρουμ κοινωνικής πολιτικής. Αυτό σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάποια επιρροή εκεί, ε, αλλά αυτή τη στιγμή δεν είναι αυτό το φόρουμ για συζήτηση τέτοιων θεμάτων. Ε, θα επανέλθω όμως και στους δύο αυτούς φορείς αργότερα. Η τρίτη διάσταση είναι η κάθετη συνοχή. εννοούμε τη σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, προς άλλες τρίτες χώρες. Ε, ο Μάικλ μίλησε για τα ήπια μέσα που έχουμε, αλλά έχουμε και κάποια άλλα πιο δεσμευτικά μέτρα. Ε, έχουμε και το GSP Plus που είναι δεσμευτικό μέσο. Υπάρχει δηλαδή ο κίνδυνο υποβάθμιση των ε, μέσων αυτών. Κατά την αξιολόγηση των μέσων, ε, ένα από τα βασικά ευρήματα είναι ότι στις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, βλέπουμε ότι η επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται με τρόπο που μοιάζει με ομόκεντρους κύκλους. Αν εξετάσουμε τις ε, χώρες της προσχώρησης ε, ή αυτές που έχουν κάποια προοπτική προσχώρησης, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρηση η αρκετά σημαντική επιρροή. Αν προχωρήσουμε πιο έξω, στον επόμενο κύκλο, ε, Φτάνουμε στις γειτονικές χώρες ε, χωρίς ε, άμεση προοπτική προσχώρησης ε, ή τις αναδυόμενες οικονομίες που είναι ο κύκλος που απέχει περισσότερο από το κέντρο. η τις αναδυομενες οικονομιες που ειναι ο κυκλος που απεχει περισσοτερο απο το κεντρο τυπολογία των χωρών που εξετάσαμε φαίνεται στην ε, σχετική διαφάνεια. Θα σας αναφέρω όμως κάποιες γενικές παρατηρήσεις προτού ε, προχωρήσω βαθύτερα στην ανάλυση των διαφόρων μέσων. Σε παγκόσμια κλίμακα βλέπουμε να υπάρχει μια δυναμική σχέση ανάμεσα στα, στα κοινωνικά πρότυπα και την οικονομική ανάπτυξη. Τα δύο πράγματα αυτά πάνε χέρι-χέρι. Και είναι σημαντικό να το έχουμε αυτό κατά νου. Ένας από τους βασικούς φορείς είναι οι πολυεθνικές εταιρείες. Είναι σημαντικοί παράγοντες στις αντιόμενες οικονομίες και ως εργοδότες, αλλά και ως κεντρικοί πολιτικοί παράγοντες, διότι έχουμε δει ότι επιχειρήσεις μέτρα την Ευρώπη προσπαθούν να επηρεάσουν ε, το εργασιακό δίκαιο σε κάποιες αναδιόμενες οικονομίες ε, όπου ουσιαστικά επιδιώκουν το αντίθετο από αυτό που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε κατά νου τον κεντρικό ρόλο των πολυεθνικών αυτών εταιριών. Μια άλλη γενική παρατήρηση είναι ότι οι αναδυόμενες οικονομίες εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από ε, τα πλεονεκτήματά τους όσον αφορά το ε, εργατικό κόστος και διστάζουν να υιοθετήσουν υψηλότερα πρότυπα. Um, Στην ε, διαφάνεια υπαριθμό 18 βλέπετε την, ε, τις επιπτώσεις των δεσμευτικών μέσων που έχουμε. Αναφέρθηκα ήδη στις στα σύμφωνα σύνδεσης. τα οποία είναι πολύ σημαντικά και επηρεάζουν σημαντικά τα ε, πρότυπα εργασίας. Το GSP+, Plus, το ε, Γενικό Σύστημα Προτιμήσεων, είναι σημαντικό μέσο ε, οι επιπτώσεις του όμως ε, είναι μάλλον ε, μεσαίας τάξης. Θα ήθελα επίσης ε, να ξαναναφέρω τον ΠΟΕ. Σημαντικό είναι να θυμόμαστε ότι πρόκειται για οργάνωση που έχει να κάνει με το εμπόριο. Θα ήταν όμως σημαντικό να συζητήσουμε πώς μπορεί να παίξει κεντρικό ρόλο στο μέλλον. Όσον αφορά τα πιο ήπια μέσα που έχουμε, τα μη δεσμευτικά, αυτή τη στιγμή οι επιπτώσεις τους είναι μεσαίου μεγέθους. Βλέπουμε ότι κάποιες χώρες αλλάζουν τακτική. Άλλο σημαντικό μέσο εδώ είναι η εταιρική ευθύνη, το οποίο συνδέεται με αυτό που είπα νωρίτερα. Συνδέεται δηλαδή με το σημαντικό ρόλο των πολυεθνικών εταιριών. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα για σημαντικές επιπτώσεις. Προς το παρόν όμως οι επιπτώσεις είναι μάλλον περιορισμένες για διάφορους λόγους τους οποίους θα επανέλθουμε. ο ορισμός δεν είναι πολύ σαφής και δημιουργεί προβλήματα, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό αργότερα. Θα ήθελα επίσης να αναφέρω τις επιπτώσεις των ε, προγραμμάτων αξιοπρεπούς εργασίας, ε, που είναι ένα σύστημα του ILO, του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας, ε, συνδέεται με την τεχνική βοήθεια που παρέχει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας είδαμε ότι η δουλειά σε πρακτικό επίπεδο έχει βοηθήσει κάποιες χώρες να υιοθετήσουν υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στα οικονομικά μέσα. Βλέπουμε ότι η αναπτυξιακή βοήθεια παίζει σημαντικό ρόλο. Το θέμα είναι να συνδεθεί αυτή με τα κοινωνικά πρότυπα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εργαστεί πολύ πάνω στο θέμα αυτό. Έχουμε και την τεχνική βοήθεια, τα οικονομικά μέσα, τα οποία επίσης ε, έχουν σημαντικό αντίκτυπο. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά ευρήματα της μελέτης αυτής και θα δώσω το λόγο στον Βέρνερ που θα μιλήσει περισσότερο ε, για τις προτάσεις και τις συστάσεις που έχουμε να κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε τώρα στο τελευταίο τμήμα. Υπάρχουν πέντε ε, βασικές προτεραιότητες που νομίζω θα ενδιαφέρουν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα ήθελα να σας εξηγήσω. Uh, πέντε προτεραιότητες, ε, μια συνεκτική, ενοποιημένη και επαγγελματική προσέγγιση. Δεύτερον, οικοδόμηση μιας ε, συνολικής, ε, μιας παγκόσμιας μάλλον κοινωνικής ε, συμμαχίας. Τρίτον, αναπτύσσοντας περαιτέρω την ήπια προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έμφαση στην υλοποίηση και την εφαρμογή, θέμα που έθιξαν ήδη οι συνάδελφοι, Τέταρτον, ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και προσαρμογή των εργαλείων που ήδη υπάρχουν. Πέμπτον, ενίσχυση ε, του ρόλου ε, των εταιριών μέσω της ε, εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τα εργατικά πρότυπα και για το εργατικό δίκαιο και όλα τα συναφή ζητήματα. Νομίζω μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα μέσω της εταιρικής ευθύνης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά δρά μέσα στο θεσμικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ένας μεμονωμένος εταίρος που έρχεται σε επαφή με διεθνείς οργανισμούς. Οπότε και για τα κοινωνικά ζητήματα, για την κοινωνική διάσταση της παγκοσμιοποίησης ε, κινείται στο θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ στην ε, διεθνή αρένα άλλοι εταίροι ε, τονίζουν πολύ περισσότερο τα θέματα εμπορίου, παραδείγματος χάρη σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Λοιπόν, η πρώτη προτεραιότητα, συνεκτική και επαγγελματική προσέγγιση. Θα πρέπει να αυξηθεί η συνεκτικότητα και οριζόντια και κάθετα. Αυτό είναι σημαντικό ε, και για την αξιοπιστία και για να έχουμε θετικέ επιπτώσεις σε χώρες μη μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Θα πρέπει να δράμε συνεκτικό τρόπο λοιπόν η Ένωση ε, για να ενισχύσει την φήμη που έχει και τον ηγετικό της ε, ρόλο για την προάσπιση των βασικών εργατικών προτύπων. Δεύτερον, ε, η συνοχή έχει ιδιαίτερη σημασία και στις σχέσεις ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και άλλους εταίρους. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο όλους ιδιαίτερους ε, στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την νεοσυσταθήσα υπηρεσία ε, εξωτερικής δράσης που θα αναλάβει κάποιες από τις ευθύνες ε, για τις εξωτερικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας βασικός εταίρος. Ε, πρέπει νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έρχεται σε επαφή με την υπηρεσία εξωτερικής δράσης και να ακουστεί η φωνή του. Από την αξιολόγηση αντικτύπου ε, προκύπτει ότι η συνοχή έχει βαρύτητα και στις διαπραγματεύσεις στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας, στην προπαρασκευαστικό στάδιο υπάρχει συνοχή, αλλά την ώρα της ψηφοφορίας. Δεν ε, υπάρχει ομοφωνία ανάμεσα στις ε, χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά. Θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Επίσης, ε, μια πιο επαγγελματική προσέγγιση στις σχέσεις με άλλους εταίρους θα ήταν ευκταία. Χρειάζεται μια συνεκτικότερη προσέγγιση λοιπόν για να προωθήσουμε την εξωτερική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ευρωπαϊκά ε, εργατικά πρότυπα. Δεύτερη προτεραιότητα, η οικοδόμηση κοινωνικού συνασπισμού, κοινωνικής συμμαχίας. Έχει πολύ καλή φήμη ε, σε παγκόσμιο επίπεδο ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχει ηγετικό ρόλο στα κοινωνικά ζητήματα σε σχέση με άλλους εταίρους όπως η ΕΠΑ παραδείγματος χάρη που έχουν NIP ε, σκληρές και μονομερείς προσεγγίσεις για την κοινωνική πολιτική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους εταίρους που θα μπορούσε πολύ ευκολότερα να αναπτύξει, να δημιουργήσει νέους συνασπισμούς και να συνεργαστεί με χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα θα θέλαμε να τονίσουμε ότι υπάρχει δυνατότητα, ίσως και παρίσταται ανάγκη, να υπάρξει στενότερη σχέση με αναδυόμενες ασιατικές οικονομίες με την Κίνα, Φερρυπίν και άλλες χώρες. Αυτό θα ήταν ε, μια καλή κατεύθυνση για την ενίσχυση του διαλόγου και της συνεργασίας. Φυσικά ε, χρειάζεται στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων να τονίζουμε πάντοτε την κοινωνική διάσταση, κυρίως ε, όταν εκπονούμε εμπορικές πολιτικές που συχνά συνιστούν ύψιστη προτεραιότητα σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται στον τομέα αυτό. Οι σχέσεις με ε, ε, διακυβερνητικές οργανώσεις. Ε, εδώ θα πρέπει να δοθεί βάρος στους συνασπισμούς, στις συμμαχίες, στη σχέση με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Μην ξεχνάτε ότι και στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να προ... μπορείτε να προωθήσετε τα κοινωνικά ζητήματα. Βέβαια, ε, είναι δυσχερές το έργο, αλλά δεν θα πρέπει να αποκλειστεί από το κοινωνικό θεματολόγιο. Η οικοδόμηση βιώσιμων λοιπόν συνασπισμών με ασιατικές χώρες και με το δίκτυο των χωρών ε, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Ε, αυτά είναι τα στοιχεία κλειδιά. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εξωτερικές σχέσεις δεν μπορεί να δρά ως αυτόνομος ε, εταίρος, αλλά μπορεί να αναλάβει ηγετικό ρόλο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, τρίτον, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είπαμε, την τελευταία δεκαετία έχει υιοθετήσει μια ποιότερη προσέγγιση ε, και βοηθά αυτή η προσέγγιση και μπορεί να είναι και πολύ πιο αποτελεσματική ε, σε σχέση με την εφαρμογή σκληρών μέτρων μέσω εμπορικών συμφωνιών. Η ήπια προσέγγιση. Φυσικά αυτή είναι, συμπληρωματική σε σχέση με τις σκληρότερες πολιτικές και ακολουθεί την κατεύθυνση της ε, περαιτέρω υλοποίησης ε, και εφαρμογής των εργατικών πρότυπων. Η κύρωση της σύμβασης ε, του ΔΟΕ είναι ένα σημαντικό σημείο, αλλά άλλο και η επικύρωση της σύμβασης, άλλο η εφαρμογή των διατάξεών της. Η τεχνική αρρωγή είναι ένα θέμα που προκύπτει αλλά δεν είναι το μόνο. Υπάρχει η ευθύνη των εργοδοτών, των εργαζομένων, υπάρχει δυνατότητα βοήθειας μέσω εκπαίδευσης ε, που μπορεί να αναλυθεί και από εθνικές αρχές, όχι μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να υπάρξει ταυτόχρονα και παρακολούθηση της εφαρμογής των ευρωπαϊκών προτύπων. Κατόπιν, ε, αυτές οι ζώνες εξαγωγών που στις αναδυόμενες οικονομίες είναι ένα σημείο που θα πρέπει να σας απασχολήσει. Ε, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τις εξαγωγές ε, για να ε, ανυψώσουμε τα κοινωνικά πρότυπα σε αυτές τις χώρες. Uh, uh, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο θα έπρεπε να ενισχύσει αυτό το κομμάτι της τεχνικής αρρωγής γιατί ξαναλέω η υλοποίηση των μέτρων είναι σημαντικότατο κομμάτι της του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να έχει απτά αποτελέσματα. Τέταρτον, ε, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και προσαρμογή των εργαλείων. Αυτό συνδέεται με το σημείο 3. Το γενικευμένο σύστημα προτιμήσεων GSP και GSP-SYN καλύπτει κάποια κοινωνικά πρότυπα και είναι ένα από τα πλέον αποτελεσματικά εργαλεία για την προώθηση των βασικών εργατικών προτύπων στις χώρες εταίρους, αλλά ε, υπάρχει σημαντικός βαθμός μη συμμόρφωση και μη εφαρμογή των προτύπων και πάλι εδώ, όπως έλεγα προηγουμένως, θα πρέπει οι ποιότερες ε, πολιτικές να συνδυαστούν με άλλες προσπάθειες ε, στα πλαίσια της πολιτικής που ακολουθούμε, ούτως ώστε οι εργατικές ε, συνθήκες αυτές ε, να ε, εφαρμοστούν σε χώρες που δέχονται πιέσεις και από πολυεθνικές εταιρείες και από άλλες παραγωγικές μονάδες που τείνουν να παραγνωρίζουν τη σημασία όλων των κοινωνικών ζητημάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συνεχίσει στα πλαίσια των εμπορικών συμφωνίων να τονίζει το βάρος που έχουν τα εργατικά πρότυπα και τα εργατικά πρότυπα, τα κοινωνικά πρότυπα επίσης ε, θα πρέπει να ενσωματώνται σε οποιαδήποτε μορφή διαλόγου, ανταλλαγή ε, εμπειριών και τεχνικών προγραμμάτων, αλλά επίσης και στα πλαίσια της αναπτυξιακής βοήθειας ε, θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο απαιτητική σε σχέση με την τηρήση των κοινωνικών προτύπων όταν χρηματοδοτεί αναπτυξιακά προγράμματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να προωθήσει τις θέσεις του και κυρίως ε, με τις ε, νέες εξουσίες που έχει με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πέμπτον, αλλά εξίσου σημαντικό είναι η εταιρική και κοινωνική ευθύνη. Ε, ενδυνάμει μεγάλη επίπτωση μπορεί να έχει η αρχή της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης σε αυτές τις μεγάλες αλυσίδες, πολυεθνικές εταιρείες ε, που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις αναδυόμενες οικονομίες λόγω των ξένων επενδύσεων. Ε, δηλαδή οι ξένοι επενδυτές είναι και μεγάλοι εργοδότες σε αυτές τις αναδυόμενες οικονομίες και ως εκ τούτου μπορούν να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τα εργατικά πρότυπα που εφαρμόζονται σε αυτές τις χώρες. Οπότε θα εν δυνάμει θα μπορούσε να γίνει κάπως σκληρότερη, σκληρότερη η κοινωνική εταιρική ευθύνη, να μην, ε, να μην έχει τόσο εθελοντικό χαρακτήρα, να υπάρχουν ελάχιστα πρότυπα, τα πρότυπα του ΑΣΕ παραδείγματο χάρη, του ΩΣΑ, συγγνώμη, για την εταιρική κοινωνική ευθύνη, εγγυήσει σε σχέση με τις επενδύσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επιβάλλει πιο δεσμευτικές υποχρεώσεις σε πολυεθνικές εταιρείες, παραδείγματος χάρη για τις ε, εγγυήσεις, για τις επενδύσεις θα ε, μπορούσαμε να δούμε πώς ακριβώς μπορούμε να εντάξουμε τα εργατικά ε, πρότυπα στις τοπικές αλυσίδες ε, διανομής και ίσως και να επικουρήσουμε τις επιχειρήσεις μέσω των εθνικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων στην εκάστοτε χώρα, ούτως ώστε να εποπτεύουν εκείνη την εφαρμογή των κοινωνικών πρότυπων. Τέλος, θα έπρεπε να συγκροτήσουμε μια εταιρική σχέση με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ε, που παρακολουθούν ε, ασθενά ε, και άγρυπνα τις παραβιάσεις των εργατικών, των διατάξεων ως προς το, τις εργατικές συνθήκες και τα εργατικά δικαιώματα. Ξαναλέω, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να δράσει μόνο του, ε, αλλά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να παρακινήσει το Κοινοβούλιο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σκληρύνει κατά τη στάση της ε, και στην εξωτερική διάσταση ε, της πολιτικής της ε, να επιβάλλει πιο δεσμευτικές διατάξεις στις πολυεθνικές εταιρείες που εδρεύουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά έχουν και θυγατρικές σε αναδυόμενες οικονομίες. Με αυτές τις πέντε λοιπόν συστάσεις θα ήθελα να κλείσω την παρουσίαση της μελέτης μας και προσβλέπουμε στα σχόλια τις παρατηρήσεις και ερωτήσεις σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Συγγνώμη τον ε, Μικαήλ Κάντια που τον ξέχασα. Και οι τρεις λοιπόν συντάκτες της μελέτης είναι εδώ. Θέλετε κύριε Μπάρφ να ε, μιλήσετε τώρα, μετά κύριο Φάλκ. Φάλκ. Κύριος Φάλμπε μάλλον. Ευχαριστώ τους ε, συντάκτες της ε, έκθεσης, ε, της μελέτης αυτής μάλλον. Θα ήθελα να θέσω διάφορες ερωτήσεις και να κάνω και κάποια σχόλια. Αναφερθήκατε στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ε, επανειλημμένα. Εάν θέλουμε να ε, πείσουμε ε, ή μάλλον να υποδείξουμε στις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ποιο τρόπο πρέπει να συμπεριφέρονται και ποια πρότυπα κοινωνικά πρέπει να εφαρμόζονται, καλά θα κάναμε πρώτα να κοιτάξουμε την κατάσταση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα την Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρετε, υπάρχουν παραβιάσεις των προτύπων του ΔΟΕ. Ε, στην περασμένη θητεία της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ε, σχέδια οδηγιών που δεν συνάδουν με τα ε, πρότυπα του ΔΟΕ, όπως παραδείγματο χάρη η οδηγία για τα ωράρια εργασίας που το Κοινοβούλιο απέρριψε στη συνέχεια. Ξέρουμε ότι υπάρχει σύμβαση του ΔΟΕ για τον ανώτατο χρόνο εργασίας και ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, πρότεινε 65 ώρες εβδομαδιαίας εργασίας. Εγώ ε, έχω υπηρετήσει επί δεκαετία ε, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΕ, εκπροσωπούσα τα συνδικάτα και σας διαβεβαιώ πως παρατηρούσα την μειούμενη επιρροή του ΔΟΕ σε διεθνές επίπεδο δέχεται διαρκώς επιθέσεις ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας ε, και ούτως ή άλλως ε, λόγω της κρίσης επιδεινώνεται η κατάσταση σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δείτε την νομοθεσία που ενέκρινε πρόσφατα η κατασταση σε ολα τα κρατη της ευρωπαικης ενωσης δειτε την νομοθεσια που ανεκρινε προσφατα η ισπανια για τις συλλογικέ συμβάσεις, πόσο δυσμενής είναι η όρη της. Για τις, τους οργανισμούς εταίρους, θα πρέπει να ξέρετε ότι οι, οι εταιρείε, α πούμε, α πάρουμε τι εταιρείε καλύτερα, έρχονται ε, σε άμεση επαφή με τι κυβερνήσει και λένε ότι αν μα επιβάλλετε τόσο αυστηρού όρου, δεν πρόκειται να επενδύσουμε στη χώρα σα. Ε, και άρα πιέζονται οι κυβερνήσει να δεχτούν του όρου των εταιρείων. Όταν ε, διαπραγματευόμασταν για τη συμφωνία από ΕΕ, στο Σιάτλ, στη Σιγκαπούρη, οι Ομοσπονδίες Ανεξάρτητων Συνδικάτων ζήτησαν από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου να προβλέψει ότι όποιος ε, δεν εφαρμόζει τα, όλα τα άρθρα και όλες τις ερήτρες ε, των εμπορικών συμφωνιών δεν μπορεί να είναι και μέλος του ΠΟΕΜ μας αρνήθηκαν, αρνήθηκαν να μπουν στο κοινωνικό κομμάτι και μας ε, ε παρέπεμψαν στο Διεθνή Οργανισμό Εργασίας. Ε, τέλος πάντων, για να ε, κλείσω αυτό το σχόλιο, πρέπει και εμείς να συμμορφωθούμε με τα πρότυπα του ΔΟΕ πριν το ζητήσουμε από άλλες χώρες. Ε, το κοινωνικό πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δέχεται επιθέσεις στη Τσεχία, στην Ισπανία, Εκδόθηκε πρόσφατα ένα βιβλίο στο Ηνωμένο Βασίλειο που περιγράφει πολύ σωστά την κατάσταση. Οι συντάκτες της μελέτης μας μίλησαν για τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε και μας εξήγησαν ότι ε, αν είναι κάπου φτηνότερη η παραγωγή τότε αυτό ουσιαστικά ισούται με αθέμητο ανταγωνισμό. Άλλες χώρες λοιπόν παράγουν ευθυνότερα αγαθά και άρα ε, εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω αυτών των ζωνών στις οποίες αναφερθήκατε ευθυνότερα προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, ξέρετε όμως ότι για να μειωθεί το κόστος υπάρχουν οι πρακτικές όπως ε, συνθήκες δουλείας στο χώρο εργασίας Στον ε, Διεθνή Οργανισμό Εργασίας ήρθαμε αντιμέτωποι με υποθέσεις όπως ε, αυτή μιας ε, γερμανικής εταιρείας που ουσιαστικά παρεμπόθησε την ίδρυση συνδικάτων και τελικά χρειάστηκε να επικαλεστούμε τα πρότυπα του Διεθνούς ε, Οργανισμού ε, Εργασίας και ε, για να περάσω στο επόμενο θέμα, υπάρχει αυξανόμενο ποσοστό αυτοαπασχολούμενων, το οποίο δυσχεραίνει την κατάσταση. Ξέρετε, σήμερα το πρωί, να αναφερθώ και σε αυτό, δεχθήκαμε την επίσκεψη Βέλγων Υπουργών και Υφυπουργών ε, και τους ζητήσαμε να μας μιλήσουν για την UNISO ε, που είναι μια ένωση αυτοαπασχολούμενων εργαζομένων εδώ στο Βέλγιο. αλλά δεν ξέρω αν ε, η UNISO συμμετέχει στην τριμερή δομή του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Συχνά επίσης μιλάμε για την ποιότητα των ε, θέσεων απασχόλησης, αλλά ξέρετε ότι ε, πολύ συχνά ε, δημιουργούνται μόνο επισφαλείς θέσεις απασχόλησης. Ο αριθμός τους αυξάνεται διαρκώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την κοινωνική εταιρική ευθύνη, δεν συνιστά αυτό πολύ καλό εργαλείο ε, συχνά τι γινόταν. Σε μια μεγάλη χώρα υπήρχε η έδρα μιας ε, πολυεθνικής επιχείρησης ε, και υπήρχαν γενιές διαδοχικές στους, μέσα στην εταιρεία που εργάζονταν στην εταιρεία και η εταιρεία ήθελε να κάνει κάτι καλύτερο για την πόλη στην οποία είχε την έδρα της. Τώρα ε, μετατοπίζονται οι εταιρείες ε, προς την ε, Ρουμανία, προς την Τσεχία και τι γίνεται με την κοινωνική εταιρική ευθύνη και τι γίνεται με αυτή τη σκληρότερη και ποιότερη προσέγγιση στην οποία αναφερθήκατε. Ουσιαστικά δεν γίνεται τίποτα. Νομίζω ότι ε, πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά ε, το παράδειγμα το οποίο δίνουμε ε, στις τρίτες χώρες γιατί γίνονται ακόμη χειρότερα πράγματα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ συμμετείχα και στις διαπραγματεύσεις της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου στην Μπογκοτά εκεί υπάρχει φυσικά δημοκρατικό έλλειμμα, η κατάσταση είναι πάρα πολύ ε, κακή ως προς τα ε, κοινωνικά πρότυπα. Το αναγνωρίζω αυτό ότι η κατάσταση εκεί είναι χειρότερη, αλλά ε, αυτό που εννοώ με την παρέμβασή μου είναι ότι θα έπρεπε να σκεφτούμε την κατάσταση μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πριν αρχίσουμε να εξάγουμε το πρότυπό μας σε τρίτες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει περιορισμένο πεδίο δράσης Βεβαίως στην περασμένη θητεία το, Κοινοβούλιο ε, καταφέραμε ε, να απορρίψουμε μία οδηγία ε, που κατοχύρωνε χείριστες συνθήκες εργασίας παραπέμποντας στο 19ο αιώνα δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι αφήστε τους ανθρώπους να ε, εργάζονται όσες ώρες θέλουν την εβδομάδα. Τέλος πάντων θα ολοκληρώσω τώρα και θα ε, δείτε τα επιμέρους στοιχεία μέσα στην έκθεση που θα εκπονήσω. Σας ευχαριστούμε. Ο κύριος ε, Τόμας Μαν και κατόπιν ο κύριος Κρίστιανσεν. Ξέχασα την κυρία Λάμπερτ και μετά ο κύριος Μαν. Κυρία Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την ε, παρουσίασή σας. Έχω μια σειρά ερωτήσεων. Εξετάζοντας τις επιπτώσεις κάποιων από τα πιο ήπια μέσα που έχετε, θεωρήσατε ότι αυτά είναι τουλάχιστον εξίσου αποτελεσματικά με κάποια από τα πιο δεσμευτικά μέτρα θεωρείτε ότι αυτό ε, έχει να κάνει με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των ανθρώπων στα μη μέτρα. Ότι επειδή δηλαδή είναι, πιο, είναι προαιρετικά ή επειδή έχουν πιο γρήγορο αποτέλεσμα. τα αποτελέσματα είναι σημαντικότερα και δεν εννοώ οικονομικά, ε, εννοώ όσον αφορά τα πρότυπα. Θα με ενδιέφερε να μας πείτε, επειδή το Κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή αναθεωρεί το GSP+, το Σύστημα Γενικών Προτιμήσεων. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ χρήσιμη η ανταλλαγή απόψεων αυτών για την Επιτροπή Εμπορίου και την ε, Επιτροπή Απασχόλησης ε, και σίγουρα και για τις ενδιαφερόμενες χώρες. Τώρα λοιπόν που εξετάζουμε το GSP+, μήπως μπορείτε να μας πείτε τι θεωρείτε εσείς ε, μεσαίου μεγέθους επιπτώσεις τι σημαίνει δηλαδή αυτό συγκεκριμένα για τις ε, συνθήκες απασχόλησης των ε, εμπλεκομένων ανθρώπων. Τώρα βλέπουμε ότι η Σρι Λάγκα έχει αποσυρθεί από τις διαπραγματεύσεις επειδή έχει αντιρρήσεις σχετικά με τον τρόπο, με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται στην αναθεώρηση και το τι απαιτείται για αυτήν. Όταν λοιπόν ολοκληρωθεί το μέσο, τι περιμένετε. Και όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, είχαμε εδώ και χρόνια σημαντικές συζητήσεις ε, για το θέμα αυτό. Ένα από τα πράγματα που μας λένε είναι ότι εμείς ως επιχείρηση εφαρμόζουμε όλα τα πρότυπα, επιδεικνύουμε ε, περιβαλλοντική ευθύνη. Αυτό ανταγωνιστικά, ε, αυτό όσο προς τον ανταγωνισμό αποβαίνει εις βάρος μας σε σχέση με άλλες επιχειρήσεις. Τα κοινωνικά πρότυπα δηλαδή αποσπούν την προσοχή των ε, μεγάλων εταιριών και το εμπόριο είναι το πιο σημαντικό όσον αφορά τα υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα γενικά. Εσείς πώς θα απαντούσατε στο επιχείρημα αυτό. Κάποιοι από εμά νομίζω θα θέλαμε περισσότερα πυρομαχικά για να απαντάμε σε τέτοιες ερωτήσεις. Τι, εννοείτε, δηλαδή, τι, τι θεωρείτε όσον αφορά τη γνώμη ότι ε, τα πρότυπα αυτά αποσπούν την προσοχή των εταιριών και το εμπόριο είναι αυτό που έχει πραγματική σημασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Θωμασμάνο με κατόπιν ο κύριος Κρίστενσεν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω για την παρουσίαση που ακούσαμε η οποία είναι χρήσιμη ακριβώς επειδή ε, ακούσαμε ε, τις ε, θέσεις αυτές και θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Ε, δεν ακούσαμε τίποτα ούτε για τη Θεσσαλονίκη, ούτε για το Δουβλίνο, ούτε για το, το, το Ρήνο. Ε, για τις υπηρεσίες αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στο Τωρίνο νομίζω ότι έχουν γίνει πολύ σημαντικά πράγματα. Υπάρχει σαφής εξωτερική διάσταση και θέλουμε να πετύχουμε το δικό μας πρότυπο για διάφορα είδη επαγγελματικής ε, κατάρτισης να ε, υιοθετηθεί από πολλές χώρες. Κάποιες από τις χώρες αυτές έχουν γίνει μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως ε, άλλες χώρες οι οποίες δεν θέλουν να γίνουν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπουν ε, όμως ότι ο τρόπος που παρέχουμε ευκαιρίες στους νέους ανθρώπους, ο τρόπος που μορφώνονται, το πώς καταφέρνουμε την ε, ολοκλήρωση. Αυτό λοιπόν ε, βλέπουν ότι δεν το κάνουμε ε, αμυντικά αλλά θετικά και αυτό είναι ένα μοντέλο από το οποίο μπορούν να μάθουν. Το Τουρίνο, το, η Θεσσαλονίκη και το Δουβλίνο είναι τρεις από τις υπηρεσίες μας. Έχουμε περιοριστεί τώρα σε σημαντικές υπηρεσίες τις οποίες θεωρούμε σημαντικούς εταίρους εμείς εδώ στην Επιτροπή μας. Κατά τη γνώμη μου αυτό λείπει κάπως. Δεύτερη παρατήρηση, το GSP Plus, η Jean Lambert είναι πρόεδρός μας ε, στην ε, αντιπροσωπεία για την ε, Νότιο Ανατολική Ασία και εγώ είμαι αναπληρωθής της είναι απαραίτητο να ληφθούν ε, μέτρα απέναντι στις μικρές χώρες. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό απέναντι στις μεγάλες χώρες, ε, την Ινδία και την Κίνα, αλλά στην περίπτωση της Σρι υπήρχαν κάποιες τέτοιες δυνατότητες και στους τελευταίους, ε, τον τελευταίο μήνα ο ε, πρέσβης της Σρι Λάγκα, ε, όχι μόνο στην Επιτροπή αλλά και στην ε, Ολομέλεια του Κοινοβουλίου, έχει τονίσει τι ήταν σημαντικό, τι έχουν πετύχει και που, ποια είναι τα θέματα πάνω στα οποία θέλουν περαιτέρω να εργαστούν. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε εάν πάρει κανεί σοβαρά το GSP+. Ε, λέμε λοιπόν εμεί ότι δεν επιτρέπουμε παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τελεία. Έχουμε λοιπόν ένα ισχυρό δεσμευτικό μέσο και πιστεύω ότι θα είναι και αρκετά επιτυχές. Τρίτη παρατήρηση, το CSR, δηλαδή η εταιρική κοινωνική ευθύνη. Συνάδελφε Φάρμπερ, μπορώ να συμφωνήσω με την ανάλυση σας, αλλά η Τζιν έχει δίκιο. Ε, προς το παρόν, το, το ερώτημα είναι αν η, η προαιρετικότητα αυτή θα πρέπει να συνεχίσει να ισχύει ή όχι. Το θέμα είναι δηλαδή τι κάνουμε με τους δικούς μας ε, εργαζομένους, πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε τους πόρους που μας δίνει η γη. Ε, πώς μπορούμε να εκπονήσουμε κάποιους όρους. Ε, θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα προτύπων. Ε, συνεχίζουμε όμως να εντοπίζουμε προβλήματα. Η χώρα μου, η Γερμανία, έχει ένα σύστημα αξιολόγησης των προϊόντων και ε, μια κατηγορία εδώ είναι το CSR. μπορούμε ε, να πουλήσουμε τέτοια προϊόντα ή όχι. Το CSR θα πρέπει να συμπεριληφθεί σίγουρα στην νομοθεσία, ε, αλλιώς ε, δεν θα έχουμε καθόλου δημόσιους δρόμους και αυτό θα είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Ο συνάδελφος Φάρπερ έχει δίκιο. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε το μοντέλο άλλων κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Άγγελα Μέρκελ προσπάθησε με την ε, διεθνοποίηση της κοινωνικής εργασίας. Ε, είπε ότι μπορούμε να πετύχουμε να υιοθετηθούν άλλα πρότυπα ε, και πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντικός ο τομέας αυτός. Έτσι θα έχουμε ισχυρή ταυτότητα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει ευρωπαϊκός προσαρτοσμός ποιότητας. Θα ήθελα λοιπόν να συμφωνήσω με τον συνάδελφο Φάρμπρ. Παρόλα αυτά έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε σε πολλούς τομείς, ε, το γνωρίζουμε αυτό. Χαίρομαι που το κοινωνικό πρότυπο τίθεται συνέχεια στην ημερησία διάταξη και ότι μιλάμε με μία φωνή ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, πράγμα που δεν συμβαίνει πάντα, αλλά θα ήταν πολύ καλό. Ε, σήμερα το πρωί θα είδατε ότι είχαμε σημαντικούς συμβιβασμούς, ε, του οποίους μπορούμε πραγματικά να στηρίξουμε. Δεν πρόκειτο για ποίηματα, δεν λέγαμε απλά ότι θέλουμε μη έναν κάποιο συμβασμό. Όχι, ήταν μια συνοδη, συνειδητή ε, προσπάθεια. Είδαμε ότι... Η, ε, ε ότι οι συμβασμοί αυτοί άξιζαν τον κόπο. Χαίρομαι πάρα πολύ που το είδα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κρίστενσεν κατόπιν ο κύριος Κοφεράτη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τους ομιλητές για την παρουσίασή τους στο πολύ σημαντικό αυτό θέμα. Συμφωνώ με τον εισηγητή μας, τον Ρίχαρτ Φάρπερ, ότι υπάρχουν εδώ κάποιες πολύ σημαντικές προκλήσεις. Αλλά μάλλον νιώθω και τόσο περηφάνεια που είμαι Ευρωπαίος, που πιστεύω ότι θέλουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Μάλλον υπάρχουν ε, διάφορες ιδέες για το τι είδου Ευρώπη θέλουμε, αλλά νομίζω ότι εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπάρχει συμφωνία ως προς το ότι θέλουμε μια κοινωνική Ευρώπη. Τα προβλήματα προκύπτουν από το ότι δεν επενδύουμε επαρκώς στο κοινωνικό μοντέλο και σε εποχές κρίσης γίνονται περικοπές ακριβώς στο κοινωνικό πρότυπο και στο πρότυπο της αγοράς εργασίας, λίγο πολύ σε όλες τις χώρες και γι' αυτό είναι σημαντικό όπως ε, υπόθηκε, εσωτερικά να ε, μπορέσουμε να κάνουμε τις απαραίτητες ρυθμίσεις, διότι όλοι είμαστε κράτη πρόνοιας, υπάρχουν φυσικά διαφορές όσον αφορά την ε, οικονομία μας, και το κοινωνικό καθεστώς μας, αλλά είμαστε όλοι κράτη πρόνοιας. Γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε συμφωνίες, συμμαχίες. Δεν πιστεύω στα ήπια μέσα όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη, όπως πιστεύει ο Τόμας Χάν. Ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιες προϋποθέσεις, διότι μόνο οι καλύτερες επιχειρήσεις ε, συμμετέχουν ε, στο CSR και υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις που δεν ενδιαφέρονται καθόλου να βελτιώσουν την κατάσταση. Θα πρέπει λοιπόν να θεσπίσουμε κάποιες απαιτήσει για αυτούς. Θα μπορούσαμε φυσικά να επιλέξουμε να μην ε, διαλέξουμε, να μην ακολουθήσουμε αυτόν τον δρόμο. Αλλά τότε θα αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο οι συνθήκες που επικρατούν σε άλλα μέρη του κόσμου να ισχύσουν και στην Ευρώπη. Δηλαδή θα αρχίσουμε να περικόπτουμε μισθούς ε, και να ανταγωνιζόμαστε με βάση τον ε, μικρότερο κοινό παρονομαστή και δεν είναι αυτό κάτι που επιθυμούμε. Για να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς άνθρωποι και σε άλλα μέρη του κόσμου, θα πρέπει να έχουν εισόδημα από το οποίο να μπορούν να ζήσουν. Και αν δεν αρχίσουμε να έχουμε τις ίδιες απαιτήσει από τους ε, εμπορικούς μας εταίρους, τότε θα μπορούν να μας κατηγορήσουν για προτεξιονισμό. Εμένα με ενδιαφέρει λοιπόν πάρα πολύ να δημιουργήσουμε αυτές τις διάφορες συμμαχίες σε διάφορα μέρη του κόσμου και πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουν να κάνουν και με τα κοινωνικά πρότυπα και με τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Θα ήθελα να σας αφηγηθώ μια εμπειρία που έζησα στην Αγγόλα. Ε, ε, έχει να κάνει με την ε, συνεργασία και Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και είδαμε τα στάδια τους που χρησιμοποιήθηκαν στο Αφρικανικό Κύπελο τον Γενάρη και είδαμε ότι χτίζουν πόλεις για χιλιάδες ανθρώπων για να, από την Λουάντα δηλαδή ώστε να, να, να προσελκύσουν κόσμο από τη Λουάντα να πάει να μείνει σε άλλα μέρη. Μόνο Κινέζοι εργαζόντουσαν ε, στα ε, στάδια αυτά και στις διάφορες αυτές πόλεις. Ούτε ένας εργαζόμενος δεν ήταν Αφρικανός. Όλο το εργατικό δυναμικό ήταν Κινέζοι και πιστεύω ότι και εδώ θα μπορούσαμε να ορίσουμε κάπως διαφορετικά πρότυπα. Έχω ακούσει επίσης ότι υπάρχουν πλοία στην Λουάντα χρησιμοποιούν ε, εχμαλώτους ε, ε, φυλακισμένους από την Κίνα που έχουν την επιλογή είτε να πάνε στη φυλακή στην Κίνα είτε να εργαστούν στην Αγγόλα. Πιστεύω ότι η Κίνα θα μπορούσε να είναι καλός εταίρος μας, αλλά θα πρέπει να έχουμε πιο υψηλές απαιτήσει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοφεράκη. Ευχαριστώ. Και εγώ πιστεύω ότι η έκθεση που μας παρουσιάστηκε είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Εγώ ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία σύντομα και να ζητήσω μια αναλυτικότερη γνώμη από τους τρεις εισηγητές. Πρώτο, έχω την αίσθηση Λόγω της ε, κρίσης ε, που διανύουμε, που είναι μια μοναδική κρίση, δεν είχαμε ξαναδεί τέτοιο πράγμα στο παρελθόν, η διάρκεια λοιπόν αυτής της κρίσης αμφισβητεί το ίδιο μας το κοινωνικό μοντέλο. Και όλοι λίγο πολύ το αμφισβητούν. Υπάρχει από τη μια η θεωρία λιγότερο κοινωνικό κράτος ε, έχουμε τόσο καλύτερα για το οικονομικό μας σύστημα συνολικά. Από την άλλη μεριά επιτίθενται σε διάφορα βασικά σημεία αυτού του συστήματος. Ξέρουμε πολύ καλά τώρα ποιοι είναι οι ιδεολογικοί στόχοι. Το καταλαβαίνουμε και παίρνουμε τις απαραίτητες αποφάσεις. Η άλλη όμως επίθεση είναι πιο ύπουλη. Δηλαδή, συλλογικές συμβάσεις και τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις τους, η συλλογική εκπρόσωπηση και ό,τι τέλος πάντων μέσα στην κοινωνία παρουσιάζει μία συλλογική μορφή. Αυτό λοιπόν πλήττεται. Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις αλλάζουν επίσης το χαρακτήρα των εγκαταστάσεών τους πριν από, μερικούς ε, χρόν, πριν από μερικά χρόνια είχαμε μία εξειδίκευση. Δηλαδή πήγαινε η πολυεθνική σε μία χώρα και η παραγωγή της συγκεντρωνόταν σε, σε τυπικά προϊόντα εκείνης περιοχής. Προϊόντα δηλαδή στα οποία υπήρχε παράδοση σε εκείνη την περιοχή. Αλλά βέβαια οι επιχειρήσεις που κάνουν αυτή την επιλογή έπρεπε να έχουν τις ίδιες κοινωνικές προδιαγραφές. Σήμερα για να επιβιώσει αυτού του είδους το σύστημα χαμηλώνουν οι προδιαγραφές. Παίρνουν δηλαδή ως μοντέλο το χαμηλότερο επίπεδο. Αυτές οι εταιρείες επίσης δέχτηκαν και ε, ενέκριναν μάλλον και την πολιτική της κοινωνικής ευθύνης. Αλλά η κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης άμα δεν έχει δεσμευτικά στοιχεία, δηλαδή άμα φτιάχνεται μόνο με την, στην εκούσια προσχώρηση, όπου η μόνη αμφισβήτηση γίνεται από τους ίδιους που κυβερνούν την εταιρεία. Έχουμε τεράστιες ζημιές. Δείτε τι γίνεται η BP ας πούμε, η οποία έχει τεράστια κοινωνική ευθύνη. Άμα δεν περάσουμε από την εκούσια προσχώρηση, στη χρήση δηλαδή αυτού του μέσου, αλλά βάλουμε και δεσμευτικά στοιχεία, δεν θα καταφέρουμε τίποτα, γιατί τελικά είναι το ίδιο το μέσο το οποίο τελικά αυτό καταργείται. Και εγώ θα ήθελα να προσθέσω μερικά πράγματα. Η πρόκληση του κοινωνικού διαλόγου. Τώρα, στη δική μας εσωτερική ιεραρχία, το θέμα του κοινωνικού διαλόγου δεν θα έπρεπε να είναι ένα από τα πρώτα σημεία των διεκδικήσεών μας και αναγνώριση προς τα έξω. Δηλαδή, δεν θα έπρεπε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης να δίνεται το παράδειγμα. Επίσης, ο Κοφεράτη ανέφερε τον εκούσιο χαρακτήρα των κοινωνικ... της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων. Το συζητήσαμε στην Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και δεν υπάρχει ομόφωνη άποψη για το θέμα. Δηλαδή, πότε η κοινωνική ευθύνη θα γίνει κάτι το υποχρεωτικό. Πώς δηλαδή όταν εμείς αναπτύσσουμε μία ιδέα μπορούμε αυτήν την ιδέα να την ερμηνεύσουμε σε νομο, δεσμευτική νομοθεσία. Και μετά το άλλο θέμα είναι η ιεράρχηση των κανόνων. Εγώ διαπίστωσα με ικανοποίηση ότι η Εγώ λοιπόν διαπίστωσα με ιδιαίτερη ικανοποίηση την παρέμβαση της ΜΠΕΙΤΕ στο G20. Και μας λέγανε τότε ότι, και μας είχαν πει στο παρελθόν μάλλον ότι η ιεράρχηση των κανόνων Πρέπει να γίνει. Αυτό δεν αρέσει καθόλου στο Λαμί, γιατί ο λαμί κάποτε μου είχε πει ότι όχι, όλοι οι κανόνες είναι ακριβώς οι ίδιοι. Λοιπόν, οι συνάδελφοι της, ε, της ΔΟΕ έχουν άλλη άποψη γι' αυτό, για τη γεράρχηση δηλαδή, των κανόνων. Πώς το βλέπετε εσείς σε σχέση δηλαδή με τη γεράρχηση των κανόνων στα πλαίσια της ΠΟΕ. Okay, thank you very much. Um... Σας ευχαριστώ. Πολλά σχόλια και ερωτήσεις ακούσαμε. Θα αρχίσω εγώ και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Σε σχέση με αυτό που μας είπε ο εισηγητής ο κύριος Φάλμπρο, Και εμεί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συμμορφωνόμαστε στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα πρότυπα του ΔΟΕ πριν να αρχίσουμε να προσπαθούμε να εξάγουμε το πρότυπο σε τρίτες χώρες. Προφανώς, εάν εμείς οι ίδιοι ε, στο ιστορικό της Ένωσης δεν συμμορφωνόμαστε με αυτά τα πρότυπα, δεν μπορούμε να το ζητάμε από τρίτες χώρες. Υπάρχουν απαιτήσει με τις οποίες καλούμεθα να συμμορφωθούμε. Σε σχέση με τον ΠΟΕ, ακούστηκαν σχόλια στην αρχή και στο τέλος της συζήτησης. Ε, υπάρχει το θέμα των κοινωνικών προτύπων που συζητείτε στον ΠΟΕ, το γνωρίζετε όλοι. Δεν μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσα σε λίγα χρόνια. Ο ΔΟΕ έχει αναδειχθεί στον πλέον σημαντικό εταιρό για τα κοινωνικά ζητήματα των εμπορικών σχέσεων, ε, ενώ ο ΠΟΕ ασχολείται με τις εμπορικές ε, πτυχές ε, των ε, συμφωνιών. Υπάρχει αυτή η διχοτόμηση. Καλό θα ήταν να υπάρξει στενότερη συνεργασία και πάλι ανάμεσα στους δύο οργανισμούς. Κατόπιν, ε, ε, η παγκόσμια οικονομία είναι εξαιρετικά δυναμική. Ε, και θεωρούμε ότι η ενίσχυση των κοινωνικών προτύπων ε, θα μας οδηγήσει σε πιο εύραστες οικονομίες και σε ισχυρότερες εμπορικές συναλλαγές. Οπότε θα είναι θετική εξέλιξη και για τις χώρες εταίρους. Οι άμεσες ε, ξένες επενδύσεις τονώνουν το οικονομικό δυναμικό μιας χώρας καθώς και τις παγκόσμιες οικονομικές συναλλαγές. Αυτό είναι μία πρόκληση για τις αναδυόμενες ε, οικονομίες. Νομίζω ότι θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να έχουμε κάποια ελάχιστα πρότυπα τα οποία θα εφαρμόζονται. Σκληρά εργαλεία τα οποία θα συμπληρώνουμε με τεχνική αρρωγή και μηχανισμούς παρακολούθησης ούτως ώστε σταδιακά να σημειωθεί ε, αύξηση της βαρύτητας των κοινωνικών προτύπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Φυσικά δεν μπορείτε να περιμένετε να εφαρμοστούν ευρωπαϊκά πρότυπα και ευρωπαϊκά κράτη ε, πρόνοιας να αναδυθούν σε άλλα μέρη του κόσμου νυχθημερών. Σταδιακά όμως ε, θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε αύξηση των προτύπων και τήρηση των βασικών εργατικών προτύπων στις χώρες που συμμετέχουν σε διεθνή εμπορικά δίκτυα. Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα βασικό στοιχείο ε, ε, μιας πιο δεσμευτικής ε, κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, ούτως ώστε οι πολυεθνικές εταιρείες να ευθύνονται επίσης για τις εργατικές συνθήκες στη χώρα όπου γίνεται η παραγωγή εκεί όπου παραδείγματο χάρη φαίνονται τα ρούχα ή ε, φτιάχνονται παπούτσια ε, τα οποία μεταπολούν σε ευρωπαϊκές ε, αγορές. Δεν μπορούμε να ζητάμε από όλε τι επιχειρήσει να εφαρμόζουν μια ομοιόμορφη αρχή κοινωνική εταιρική ευθύνη, αλλά τουλάχιστον να υπάρχει ένα σκληρό πυρήνα ε, κοινωνικών απαιτήσεων που θα εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες λαμβάνοντας ε, υπόψη πάντοτε το ότι πολλές πολυεθνικές έχουν ε, θηγατρικές σε χώρες λίγο απομακρυσμένες από τη χώρα της έδρας. Η κοινωνική εταιρική ευθύνη δεν ε, μπορεί να ταυτιστεί με το μάρκετινγκ, ε, δηλαδή να βασίσουμε την πολιτική μας σε σχέση με τη ζήτηση στην χώρα, στη βασική χώρα δραστηριοποίησης. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κατάσταση που επικρατεί στις χώρες όπου εδρεύουν οι θηγατρικές. Τι άλλο, τι άλλο. Ο κύριος Μαν μας μίλησε για τη, τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τις υπηρεσίες. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και αυτές οι δραστηριότητες ε, και τις αναφέρουμε στην ε, μελέτη. Λέμε ότι, είναι κάτι, ότι αποτελούν μια εφικτή λύση, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορέσει να προσφέρει παραδείγματος χάρη εκπαιδευτικά σεμινάρια ε, στους τοπικούς φορείς, ε, τα, τους υπαλλήλους της δημόσιας διοίκησης ε, σε αυτά τα κράτη. Η αρρωγή είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και το τονίζουμε μέσα στην έκθεση και το άλλο σημαντικό κομμάτι είναι η υλοποίηση των μέτρων που έχουν εγκριθεί ή θα εγκριθούν. Τι άλλο, το σύστημα γενικευμένων προτιμήσεων, GSP και GSP συν και μας μας ικανοποιεί τη λειτουργία αποτελεσματικά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί με σκληρό τρόπο αν υπάρξει παραβίαση βασικών προτύπων ε, στην περίπτωση της ε, Σρι Λάγκα, νομίζω ε, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε το GSP, αλλά χρειάζεται συνοχή στην δράση μας, γιατί υπάρχουν και παιχνίδια ισχύω και άλλοι, άλλες παράμετροι που επηρεάζουν τις σχέσεις ανάμεσα στις χώρες. Ο κύριος Κομφεράτη τι μας είπε, μας μίλησε για την τωρινή κρίση. Ε, μιλήσατε για την βιωσιμότητα του κοινωνικού μοντέλου, δοθήσεις της κρίσης. Δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Ε, ξέρετε κάποιες χώρες ε, για τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης επωφελήθηκαν από την κρίση γιατί έχουν νέα νομιμοποίηση ως προς την κοινωνική προστασία και, την, ε, και ε, ε, κάποια αστάθεια που ίσως υπήρχε στο παρελθόν σταθεροποιήθηκε διορθώθηκε μέσω νέων θεσμικών δομών σε κάποιες χώρες. Δηλαδή, ε, ορισμένες φορές η κρίση είναι και ευκαιρία για να επιφέρουμε βελτιώσεις στα ευστάμινα συστήματα. Θέλετε εσείς να προσθέσετε κάτι? Θα ήθελα να προσθέσω κάποια πράγματα όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Το αν θα είναι προαιρετικό ή όχι μέτρο έχει πιο πολύ να κάνει με την παρακολούθηση και την εποπτεία. Γι' αυτό μιλάμε για χρήση των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων και των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης ε, ως θεματοφύλακης, δεν αρκεί απλά να υιοθετήσουμε ε, μια έκθεση. Είδαμε και το θέμα των εγγυήσεων για τις επενδύσεις, το οποίο συνδέεται με αυτό. Η προσπάθεια είναι να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις ώστε να επικεντρωθούν στο σύνολο της, ε, ε, της αλυσίδας παραγωγής και να διασφαλίσουν τη θέση τους και στις αναδυόμενες οικονομίες. Αυτά είναι πολύ σημαντικά ε, θέματα. Υπάρχουν πολύ καλά παραδείγματα, όπως για παράδειγμα το Ελσαλβαδόρ. Ένα από τα βασικά σημεία της μελέτης αυτής είναι η επικέντρωση στην επιβολή του νόμου, διότι είδαμε για παράδειγμα στην περίπτωση της Λευκορωσίας ότι η επιβολή του νόμου και η ε, απόσυρσή τους από το GSP Plus ε, δεν είχε τόσο τρομερά αποτελέσματα όσο ελπίζαμε. Δεν λειτουργεί λοιπόν ως ε, δεσμευτικό μέσο. Θέλαμε λοιπόν να δώσουμε κάποιες ιδέες για το πώς μπορούμε να εργαστούμε πάνω στο θέμα αυτό στο μέλλον. Η επιβολή του νόμου συνδέεται με το πώς θα γίνει και πιο διαφανές το μέσο, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να εργαστούμε πάνω αυτό στα πλαίσια του GSP. Και επίσης όσον αφορά την ε, κοινωνική συμμαχία, η Κίνα θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα. Είναι σημαντικό αυτό που κάνει η Κίνα αυτή τη στιγμή διευρύνει το ρόλο τη όσον αφορά τις άμεσες ε, επενδύσεις. Κατά κάποιο τρόπο θα μπορούσε να θεωρήσει κανεί ότι εξάγει χαμηλότερα κοινωνικά πρότυπα και ναι αυτό είναι πρόβλημα. Έχουμε για παράδειγμα το, ε, την περίπτωση της Βυρμανίας. Ε, θα πρέπει να τα γνωρίζουμε αυτά. Η δημιουργία κοινωνική συμμαχία με την Κίνα θα έπρεπε να είναι σημαντικό θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Πολύ ωραία. Ήταν ε, πληρέστατες οι απαντήσει σας μετά από αυτή την πρώτη συζήτηση για τη μελέτη σας. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε σε αυτή τη μελέτη όταν θα εξετάσουμε την έκθεση του συναδέλφου ε, Ρίτσαρντ Φάλμπρε. Πρέπει να πάω διακοπές γιατί παραμιλάω, λέει η Πρόεδρος. À σας ευχαριστούμε λοιπόν και φτάνουμε τώρα ε, στο τελευταίο σημείο της ημερησίας διατάξεως για την ε, εξέταση των τροπολογιών για την έκθεση του κυρίου Τόμα Σεμάνη για τη δημογραφική πρόκληση και για την ε, αλληλεγγύη ανάμεσα στις γενναίες. 253 τροπολογίες έχετε λάβει κύριε Σιγητά. Ε, φαντάζομαι ότι δεν θα τις σχολιάσετε μία-μία. Παρακαλώ, συνοπτικά, συνοπτικά ε, σκιαγραφίστε την συνολικότερη προσέγγιση για αυτές τις ε, τροπολογίες. Ο κύριος Τόμας Μάν, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα δούμε, θα δούμε, θα το προσπαθήσω και θα δούμε. Θα κάνουμε τεστ, αν τα καταφέρνω. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τους ε, συναδέλφους για τις πολλές τροπολογίες. 253 ε, ε, οι πολιτικές ομάδες εκπροσωπούνται σημαντικά. Είναι λοιπόν ένα θέμα που έχει απασχολήσει όλους μας πολύ. Διαπίστωσα ότι υπήρχαν πολλές τροπολογίες οι οποίες θεωρώ ότι εμπλουτίζουν το κείμενο. Από τις πολλές αυτές τροπολογίες έχω εκπονήσει 30 συμβαστικές ε, τροπολογίες. Ε, δεν κατάφερα να τις ε, στείλω όλες, διότι ήθελα μετά τη σημερινή συνεδρίαση να συνενοηθώ με τους συναδέρφους. Κατόπιν έχουμε το, τις ερνές διακοπές. Ήθελα όμως να ε, στείλω στα αγγλικά και στα γερμανικά ό,τι έχω αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι αυτό θα είναι αρκετό για να δούμε σε τι βαθμό ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους συμβασμούς αυτούς ε, και κατόπιν θα δούμε ποια θέματα θα, μπορέσουν, θα μπορέσουν να βρουν τη συμφωνία μας και ποια όχι. Κάποιες διατυπώσεις ήταν πολύ ενδιαφέρουσες. Προσπάθησα Πάντα προσπαθώ να έχω σύντομες εκθέσεις. Κάποιες ε, πολύ καλές ε, σκέψεις υποβλήθηκαν, ίσως θα μπορούσαμε στους ε, συμβιβασμούς να τα συνοψίσουμε αυτά για να είμαστε πιο επικεντρωμένοι. Θα ήθελα καταρχήν να αναφέρω το ΕΡΚ, διότι έχει κάνει έχει υποβάλει τις περισσότερες τροπολογίες, 75 ε, τροπολογίες. Ε, για τρεις τροπολογίες έχω ερωτηματικά. Θα ήθελα να τις εξετάσω με τους συναδέλφους μας. Ε, και για, μία τροπολογία δεν μπορώ καθόλου να συμφωνήσω, αλλά νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε διμερώς. Η δεύτερη ομάδα είναι η Άλτε, η Φιλελεύθερη. Ε, χαίρομαι που έχουμε εδώ κάποιους φιλελεύθερους μαζί μας. 50 τροπολογίες, ε, ε, με τις 35 ε, μπορώ να συμφωνήσω, η Λίσλιν έχει υποβάλει μόνη τις 30. Βρίσκω ότι είναι πολύ ε, καλές, αναφέρουν την ε, προοπτική των νέων μαζί με τους πιο ηλικιωμένους. την 24 Τροπολογίες από τις 30 έχουν το OK από μένα. Συμφωνώ και με άλλες τροπολογίες, 7 τροπολογίες, ε, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω, θα τα λάβετε αυτά γραπτά. Ε, θα ήθελα να συμπεριλάβω και αυτές στους συμβασμούς και ε, μία από τις τροπολογίες θα ήθελα να την υιοθετήσω όσο έχει. Πρόβλημα έχουμε τέσσερις τροπολογίες, την 69, την 200, την 239, και την 169. Ε, θα πρέπει να υπάρξουν νέες ε, νομοθετικές ρυθμίσεις ε, για κατά τη διάκριση των ηλικιωμένων. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται αυτό. Δεν χρειάζονται νομοθετικά μέτρα. Εγώ θα χαιρόμουν εάν με τις ρυθμίσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, εάν θα μπορούσαν τα κράτη-μέρη να τηρήσουν αυτά για τα οποία έχουν δεσμευτεί μέχρι στιγμής. 19 και 20 είναι τροπολογίες τις οποίες δεν μπορώ να δεχτώ γενικά. Ε, με κάποιες μικρές διορθώσεις όμως ε, γενικά μπορούμε ε, νομίζω να συμφωνήσουμε. Η κυρία Χάρκιν έχει υποβάλει τέσσερις τροπολογίες συμφωνώ, η συναδελφός από τη Γερμανία, έχω ερωτηματικά σε δύο, έχει υποβάλει πέντε τροπολογίες συνολικά με τις οποίες μπορώ να συμφωνήσω. Ο κύριος Κάτσινα από την Σλοβενία, έχω πρόβλημα με την ε, τροπολογία σας υπαριθμών 46, διότι λέει ότι ε, θα πρέπει να έχουμε μια κατάσταση ότι δεν θα πρέπει να ε, διατυπώσουμε μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν όλοι. Ε, με αυτό διαφωνώ. Εγώ πιστεύω ότι ε, θα είναι καλό να έχουμε μια κατάσταση από την οποία κερδίζουν όλοι. Θα πρέπει να επωφεληθούν και οι νέοι και οι ηλικιωμένοι από την κατάσταση αυτή. Αλλά θα μπορούσαμε ίσως να το συζητήσουμε αυτό. Η κυρία Οβίρ έχει υποβάλει έξι τροπολογίες. Ε, πρόβλημα έχω με την 206, διότι λέει ότι ε, κατά τη γνώμη μας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να παίξει συντονιστικό ρόλο στον τομέα της υγείας. Ε, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να παίξει σημαντικό ρόλο η Ευρωπαϊκή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται σε όλο. Όσον αφορά τους ε, ε σοσιαλδημοκράτε, 48 τροπολογίες, μπορεί να συμφωνήσω με 34. Για με 6 τροπολογίε έχω πρόβλημα συνάδελφος ε, Φρανσουάς Καστέξ. Ε, ε, έχουμε συνεργαστεί σε πολλές τροπολογίες. Μπορώ να συμφωνήσω με όλες τις τροπολογίες εκτός από δύο, όπου έχω μια ερώτηση. Και μάλιστα στο σημείο 17, εγώ θέλω κίνητρα για τους ανθρώπους άνω των 60 για να βρουν εργασίες. Αυτό θέλεις εσύ να το διαγράψουμε. Ε, εμείς θέλουμε να αυξήσουμε την απασχόληση των ε, ηλικιωμένων ε, στις περιπτώσεις όπου μπορούν να εργαστούν. Κάποιος που θέλει και μπορεί να εργαστεί θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να εργαστεί. Πολύ συχνά βλέπουμε ότι λέμε στους ηλικιωμένους ότι είσαστε μεγάλης ηλικίας. Αυτό βρίσκω ότι είναι διάκριση. Ε, αυτό είναι το ένα σημείο και το άλλο είναι η τροπολογία 167 που έχει να κάνει με το όριο ηλικίας για την ε, συνταξιοδότηση. Ε, βρίσκω λάθος μία ε, διευκρίνηση ανατομέα. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μια ευέλικτη λύση και όχι μια ενιαία λύση. Μπορεί να διαφωνούμε εδώ πέρα, αλλά πολύ ευχαρίστως να το συζητήσουμε αυτό. Δέκα τροπολογίες από την ε, Χωβάνα Πάπλας ε, μπορώ να συμφωνήσω σχεδόν με όλες. Πρόβλημα έχω μόνο με το σημείο 17 που έχει να κάνει με την βαθμία κατάργηση της ε, πρόορης σύνταξης. Στη Γερμανία προσπαθήσαμε να πετύχουμε την πρόορη σύνταξη για να ε, δώσουμε περισσότερες ευκαιρίες ε, στους νέους. Ε, αλλά το δεύτερο μέρος ε, του σχεδίου αυτού δεν ε, εφαρμόστηκε, δηλαδή ε, σταμάτησαν πολύ να εργάζονται χωρίς να δίδονται ευκαιρίες στους νεότερους. Αλλά γενικά βρίσκω ότι είναι πολύ λάθος το μήνυμα ότι α, είστε πολύ μεγάλος να φύγετε από τη δουλειά. Με, η κυρία Ράπτη έχει υποβάλει τροπολογίες, έχω πρόβλημα με την εγγύηση για τους νέους, αλλά το το εξάμεινο έχει περιοριστεί εδώ σε τετράμινο. Για κάποια κράτη-μέλη πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν είναι καθόλου ρεαλιστικό. Εάν έχουμε έξι μήνες ε, για να δώσουμε στους νέους τη δυνατότητα να λάβουν μια θέση απασχόλησης ε, ή μια πρόσθετη κατάρτιση ή συνδυασμό αυτών των δύο, ε, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε προχωρήσει σημαντικά. Η κυρία Ζίπελ από τη Γερμανία έχει υποβάλει τέσσερις τροπολογίες Συμφωνώ με όλες εκτός από την 83, διότι είπε ότι οι πτυχές ασφαλείας θα πρέπει να εξεταστούν περισσότερο από ότι η ευελιξία. Εγώ είμαι υπέρ ισορροπίας μεταξύ των δύο. Ε, ο, ο Λε Κρίστενσεν έχει υποβάλει τροπολογίες. Όλε ξέρεις πάντα ότι σε υποστήριξα. Ε, ε δεν θα ε, ζητήσω τροποποίηση. Η συνάδελφος από την Λιθουανία των Σοσιαλδημοκρατικών έχει υποβάλει 8 τροπολογίες συμφωνώ με όλους. Το ίδιο ισχύει για την κυρία Κλειτή από τη Ρουμανία όσον αφορά τους, ε, την ΚΟΕ. 45 τροπολογίες έχουν ε, ε, υποβάλει, με τις 13 τροπολογίες έχω πρόβλημα. Η κυρία σήμερα έχει υποβάλει πέντε, συμφωνώ απόλυτα. Μία ερώτηση έχω όσον αφορά την, τον περιορισμό του χρόνου εργασία. Θέλετε διεύρυνση στον τομέα των δημοσίων υπηρεσιών λόγω τη ε, δημογραφική ε, ε, μεταβολή. Δεν συμφωνώ με αυτό. Ο πατρική Ριάκα από τη Γαλλία έχει υποβάλει 35 τροπολογίε. Μπορώ να συμφωνήσω με τι 10 και με την 166 μπορεί να συμφωνήσει τη φροντίδα των ηλικιωμένων, αλλά ζήτησε αύξηση της φορολογίας. Ε, υποστηρίζει την πρόορη σύνταξη στην 127 ε, και θέλει και... Ε, εγώ θέλω ευελιξία, δεν θέλω μια ενία λύση. Ο κύριος Χίγκινς έχει υποβάλει 14 τροπολογίες. Το μόνο με μία έχω σημαντικό πρόβλημα, την 41 ε, θέλει την ε, η οικογένεια ως ε, βάση της κοινωνίας δεν μπορώ να συμφωνήσω με κάτι τέτοιο. Σήμερα είχαμε συζήτηση με την οποία δεν μπορούσα καθόλου να συμφωνήσω και όσον αφορά την μείωση της εβδομάδας εργασίας διαφωνώ. Όσον αφορά τους πράσινους, 22 τροπολογίες έχουν υποβάλει, η κυρία Κορνέλησεν ε, τις έχει υποβάλει, με τις 16 μπορώ να συμφωνήσω και τις βρίσκω πολύ καλές, έχω όμως πρόβλημα με το τετράμινο της εγγύησης των νέων, εγώ ήθελα 6 μήνες, ε, το είπα αυτό και πριν. Σημαντικό βρίσκω να προωθούμε αλλά και να απαιτούμε και στο 32 θέλουμε επιτυχή ε, ένταξη και γι' αυτό θέλουμε ε, συνεργασία και από τις δύο πλευρές διότι θα πρέπει να είμαστε διατεθειμένοι να πετύχουμε την ε, ένταξη. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Έχουμε πρόβλημα με αυτό. Έχουμε πρόβλημα και με την οδηγία πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, σήμερα κατά την ψηφοφορία της έκθεσης του συναδέλφου Χέντελ ε, είχαμε το θέμα αυτό, δεν συμφωνήσαμε, αλλά πιστεύω, βρήκαμε συμβιβασμό στην έκθεση του συναδέλφου Χέντελ και Τέλος, ε, έχουμε το ECR. Ε, ε, ο συνάδελφος είναι εδώ, έχει υποβάλει πολλές τροπολογίες. Μπορώ να συμφωνήσω με τις έξι από αυτές. Με τις άλλες έξι έχω λίγο πρόβλημα. Αναφέρεις, για παράδειγμα, τη φροντίδα των μικρών παιδιών Ε, αμφισβητείς ε, αυτά που είναι για μένα εμπειρίες από τη δική μου χώρα. μπορώ να το συζητήσουμε αυτό. Ε, αλλά μπορώ να συμπεριλάβω κάποια μέρη των τροπολογιών σου στις συμβαστικές τροπολογίες. Συμφωνώ με πολύ μεγάλο μέρος των τροπολογιών. Έχω κάποια προβλήματα με κάποιες τροπολογίες, ε, αλλά είμαι διατεθειμένος ε, και κάποια σημεία να τα συμπεριλάβω σε συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Euh, ευχαριστώ κύριε εισηγητά. Η κυρία Λιν. Μάλιστα. Ε, ευχαριστώ που μιλήσατε για τις τροπολογίες μου από διαδικαστική πλευράς όταν θα συνθέσετε τις ε, συμβαστικές τροπολογίες γιατί κάποιοι θα αποχωρήσουν αύριο το πρωί. Ξέρω ε, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της έκθεσης αλλά ήθελα να πω όταν θα, ε, θα θελήσετε πότε θα διαπραγματευτείτε τις συμβαστικές τροπολογίες με τους συναδέλφους. Εγώ θα φύγω αύριο για το Ηνωμένο Βασίλειο. Μήπω μπορείτε να μα στείλετε email τις επόμενε ημέρες. Ε, τώρα, επί της ουσίας, είπατε ότι δεν ε, θα μπορέσετε να συμφωνήσετε με όλες τις τροπολογίες μου. Κάποιες δεν σας βρίσκουν σύμφωνο, το φανταζόμουν. Ε, πρέπει να εφαρμόζουμε την εγκεκριμένη νομοθεσία, λέω σε μια τροπολογία μου. Οπότε, συμφωνείτε με τις τροπολογίες που σχετίζονται με αυτή την αρχή. Υποθέτω ναι. Για την νέα οδηγία που εξετάζεται από το Συμβούλιο τώρα. Ε, υποθέτω ότι θα μιλήσουμε για τις δημογραφικές προκλήσεις και δύσκολα μπορούμε να αναφερθούμε σε αυτές, χωρίς να ε, παραπέμψουμε για, στην καθολική πρόσβαση υπηρεσίες ε, και στην κατάργηση της διακριτικής μεταχείρισης. Γι' αυτό υπέβαλα εγώ τις για τροπολογίες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενέχει και αυτό το σημείο ε, η έκθεση, γιατί έχουμε το πακέτο του άρθρου 13 και πάντοτε προκύπτουν τα ίδια προβλήματα. Δεν έχει καμία σχέση με την απασχόληση, μιλάμε για πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και μόνο. Ελπίζω να βρούμε κάποιο σημείο συμφωνία χωρί να χρειαστεί να αποσύρω τι τροπολογίε. Ξέρω, ξέρω ότι έχετε κατά νου αλλά ελπίζω να βρούμε μια άλλη λύση. Ε, γιατί η οδηγία για την ε, καταπολέμηση της διακριτικής μεταχείρισης ε, θα υπάρχει πρόβλημα με όλους τους βουλευτές από τη Γερμανία. Δηλαδή στη Γερμανία πώ θα πείσετε ότι θα πρέπει να εξαχθεί το γερμανικό μοντέλο σε άλλες χώρες, να εφαρμοστούν οι ίδιες διατάξεις σε άλλες χώρες. Μα εσείς δεν καταλαβαίνω γιατί αγωνίζονται οι Γερμανοί βουλευτές, ενώ στη Γερμανία ήδη ισχύουν αυτές οι διατάξεις. Ε, τώρα, σχετικά με την υποχρεωτική ε, ηλικία συνταξιοδότησης ε, θα συμφωνήσω, αλλά ας μιλήσουμε για ευέλικτη ηλικία συνταξιοδότηση καλύτερα, γιατί δεν θα πρέπει να μπορεί ο εργοδότης να υποχρεώνει κάποιον να συνταξιοδοτηθεί εφόσον έχει τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα και εφόσον προβλέπεται η χορήγηση της σύνταξης από κάποια ηλικία και μετά. Ε, κατόπιν πρώτη να τροποποιήσει της ε, παραγράφου 11 γιατί φαίνεται σαν να λέτε ότι η ευελιξία ε, και ασφάλεια στις προσωρινές θέσει απασχόληση είναι ένα εμπόδιο. Ξέρετε, σε ορισμένε περιπτώσεις κάποιοι πιο ηλικιωμένοι θέλουν να δουλεύουν μόνο μία-δύο ημέρες την εβδομάδα. Δεν θέλουν απαραίτητα να έχουν πλήρη απασχόληση. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα μηχανισμό που θα εξετάσουν τα κράτη-μέλη, να εξετάσουν και αυτήν την εναλλακτική λύση τη ευελιξία να κάποιοι, αν δηλαδή ο εργαζόμενο θέλει να, μια μερική απασχόληση, να έχει και αυτή την επιλογή. Ε, ανταλλαγή των πρακτικών. Καλό θα ήταν ε, να αυξηθεί ε, για την φροντίδα των συγγενών. Δηλαδή, πολλοί δεν έχουν συγγενείς, αλλά δεν θέλουν παραδείγματο χάρη να πάνε σε κάποιο οικοευγυρία, σε Γι' αυτό και υπέβαλα μια τροπολογία. Καλό θα ήταν να γίνει ανταλλαγή ε, ε, εμπειριών ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Δηλαδή τι θα κάνουμε ε, με τους ανθρώπους που δεν θέλουν να μπουν σε κάποιο ίδρυμα παρότι δεν έχουν συγγενείς. Και καλό θα ήταν οι ηλικιωμένοι να έχουν πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους σε προσβάσιμο μορφότυπο, δηλαδή το ίδιο ισχύει και για τα άτομα με αναπηρίες. Ε, νομίζω ότι όλα θα πρέπει, όλες οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσβάσιμες για όλες τις ε, πληθυσμιακές ομάδες. Σε κάτι άλλο, μιλήσατε για την περίθαλψη. Ωραία, εγώ θέλω να διευρύνω αυτό που είπατε στην υγειονομική περίθαλψη. Ξέρω ότι δεν υπάρχει αρμοδιότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλω να αλλάξει. Ε, δεν θέλω να αλλάξει απαραίτητα αυτό, αλλά κάποιε πτυχέ τι καλύπτουμε στην υγειονομική περίθαλψη και θα ήταν σημαντικό να δούμε τι ε, εθνικές ε, παραδόσεις και να διαπιστώσουμε ότι κάποιοι δεν έχουν πρόσβαση σε συγκεκριμένα φάρμακα, παραδείγματο χάρη. Ε, καλό θα ήταν τα κράτη-μέλη να γνωρίζουν ότι μας απασχολεί ε, αυτό το θέμα. Κάποιοι δηλαδή που δεν έχουν πρόσβαση σε φάρμακα λόγω ηλικίας, παρότι νοσούν. Ε, θα υποβάλω και την προφορική ερώτηση και την πρόταση ψηφίσματος. Ξέρω ότι το αναφέρατε αυτό στην έκθεσή σας, γιατί έχουμε συνεργαστεί από αυτό στο παρελθόν. Ελπίζω να ε, δεχτείτε τα περισσότερα από αυτά τα σημεία, παρότι έχετε κάποιες επιφυλάξεις ε, για τη διακριτική μεταχείριση. κυρία Καστέξ, τώρα λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για τις ε, προσπάθειες συμβιβασμού που φαίνεται να κάνει. Βέβαια είναι δύσκολο να, να συμφωνήσουμε όταν δεν το έχουμε μπροστά μας γραπτά αυτό το οποίο προτείνεται ως συμβιβασμό. Εγώ θα ήθελα να σας πω ε, για τους σοσιαλιστές θα υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές πάνω στις οποίες εμείς θα βασιστούμε και όρια να μην ξεπεράσουμε. Δηλαδή να έχουμε μία νόμιμη ηλικία αναχώρησης ε, για σύνταξη, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε όμως να έχουμε και μία ψαλίδα ηλικίας διότι το ποσό της σύνταξης που πρέπει να διασφαλίζει αξιοπρεπή γεράματα εξαρτάται από την νόμιμη ηλικία αποχώρησης. Τώρα βέβαια με την παράταση του ανθρωπίνου βίου σίγουρα χρειάζεται και η αντίστοιχη περίοδος εισφορών για την Flexi Security θέλουμε το κοινωνικό στάνταρ να είναι εγγυημένο και θέλουμε επίσης για εκείνους οι οποίοι εναλλάσσουν απασχόληση με κατάρτιση, θέλουμε η κατάρτιση να μετριέται ως συντάξιμη ηλικία. Αυτό μπορεί να εξαρτάται από τη μία χώρα στην άλλη. Μπορεί να είναι 39, μπορεί να είναι 42 χρόνια. Θα πρέπει τουλάχιστον όμως να έχουμε αυτά τα 40 χρόνια ενεργού βίου που πρέπει να διασφαλίζουν την αξιοπρεπή σύνταξη και δεν πρέπει μόνο στα γεράματα να ρυθμίζονται αυτά τα πράγματα αλλά σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ζωής πρέπει να προβλέπεται η αποχώρηση στη σύνταξη. Εμείς θέλουμε όταν γίνεται διαφοροποίηση ανάλογα με τον κλάδο να λαμβάνεται υπόψη και η βαρύτητα της δουλειάς, η φύση της δουλειάς και η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων έχει ξεκινήσει κλαδικές ε, συνομιλίες σχετικά, διότι υπάρχουν δουλειές ιδιαίτερα βαριές και κουραστικές που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποχώρηση στην σύνταξη. Αυτά είχα να πω και μετά θα δούμε με τις συμβιβαστικές τροπολογίες άμα θα πρέπει να συνεχίσουμε ή όχι τη συζήτηση. Ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που αργήσα. Ήμουνα σε συνεδρίαση άλλης επιτροπής. Η κυρία ημουνα σε συνεδριαση αλλες επιτροπης η κυρια λαμπερτ ε, μου μετέφερε κάποια από τα σχόλιά σας για τις τροπολογίες μας. Είναι πολύ θετικό βρίσκο που ε, προτίθεστε να ενσωματώσετε πολλά από τα σχόλιά μας ε, στην έκθεσή σας. Ε, πραγματικά είναι σημαντικό που τονίζετε ότι σχετίζεται με την ισότητα των δύο φύλων και σήμερα στην Επιτροπή Γυναικών ψηφίσαμε και την έκθεση της κυρίας Μπάουερ και θα σας τη διαβάσουμε προφανώς. Θα ήθελα τώρα εν συντομία να σας πω κάποια πράγματα για την εγγύηση για τους νέους. Είπατε ότι προτιμάτε ε, τους έξι μήνες που προτείνετε εσείς και όχι τους τέσσερις που προτείναμε εμείς. Πλην όμως ε, τον περασμένο μήνα στην Ολομέλεια ε, ψηφίστηκε η έκθεση της κυρίας ε, σχετικά και ξέρετε ε, το, το, σώμα, το κοινοβούλιο έχει ψηφίσει ήδη τους τέσσερις μήνες. Ε, θα ήταν πάρα πολύ παράξενο λοιπόν τώρα να είπα να χωρίσουμε γιατί ήδη σε μια άλλη έκθεση έχουμε προτείνει ε, τους τέσσερις μήνες και έχει ήδη ψηφιστεί η έκθεση έκθεση. Ε, τώρα για την τροπολογία 21 σχετικά με την ε, διπλή ένταξη, την, ε, την ε, προσέγγιση σχετικά με την ένταξη, συμφωνούμε ότι πρέπει να είναι δυσδιάστατη. Ε, αυτό αναφέρεται στην πρώτη πρόταση, αλλά εμείς προτείναμε να διαγραφεί το κομμάτι που ε, βαρύνει περισσότερο ε, τους νέους εισερχόμενους σε σχέση με αυτούς που ήδη είναι εκεί. Δηλαδή λέτε ότι οι μετανάστες πρέπει να προσαρμοστούν και όχι η κοινωνία που τους υποδέχεται. Ξέρετε ότι κατά τη γνώμη μου ε, υπάρχει πολύ καλύτερη ισορροπία αν χρησιμοποιήσουμε την ε, διατύπωση της ε, πρώτης αράδας, να ρίξουμε βάρος στην πρώτη αράδα της παραγράφου. Είναι πολύ πιο ισορροπημένη. Αυτά λοιπόν και μετά το, ε, τις καλοκαιρινές διακοπές θα συζητήσουμε και πάλι τις τροπολογίες. Ε, η κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ. Ένα σύντομο σχόλιο. Ε, ευχαριστώ ε, τον εισηγητή. Έκανε πολύ θετικά σχόλια για τις τροπολογίες που έχω υποβάλει. Ζητώ συγγνώμη γιατί μπήκα στην αίθουσα αμέσως μετά την παρέμβασή σας όπου μιλούσατε για τις τροπολογίες μου. Με ενημέρωσε όμως κυρία Λάμπερ. Τέλος πάντων, το μόνο που θέλω να πω σχετίζεται με το, αυτά που είπε ο συνάδελφος από τους σοσιαλιστές, αλλά δεν είναι ταυτόσιμο το σχόλιο. Οι 48. Εκεί μιλάω για το συνδυασμό της ε, αμοιβή απασχόλησης ε, και την κοινωνική ασφάλιση. Δηλαδή τι εννοώ. Ε, αυτοί που θα πρέπει να φροντίσουν κάποιον και πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται άνευ οπαδοχών θα πρέπει να καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση ούτω ώστε να μην έχουν χαμηλότερη σύνταξη στο τέλος όταν φτάσουν ηλικία συνταξιότητες, επειδή διέκοψαν για μια περίοδο για να φροντίσουν κάποιο συγγενή. Γι' αυτό σας λέω σχετίζεται με το σχόλιο τη αδέλφια από τους σοσιαλιστές ε, που έλεγε ε, ότι ζητώ συγγνώμη, διορθώνει ο μιλήτριο, Είπατε εσείς ε, να μην χάσει κάποιους παροχές, να μπορεί ο ίδιος να καταβάλει τις αντίστοιχες εισφορές κατά την περίοδο που διακόπτει την αποσχόλησή του, να πληρώνει τις εισφορές στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Πρόεδρος, υπάρχει κάποιος άλλος, όχι, τότε θα δώσω το λόγο στον εισηγητή για να κλείσουμε και τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Θα είμαι σύντομος. Κυρία Λίν, πολλούς συμβιβασμούς έχουμε πετύχει στο παρελθόν. Σίγουρα θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. Όσον αφορά τις ε, διακρίσεις, ε, δεν, έχουν, δεν έχει αλλάξει η κατάσταση, όχι μόνο όσον αφορά μας τους δύο, αλλά και άλλους. Μέχρι αύριο το απόγευμα θα προσπαθήσω να έχω τις ε, συμβαστικές προτάσεις ώστε να μπορώ να σας τις στείλω. Στην πρώτη εβδομάδα μετά τις ε, θερινές διακοπές θα μπορέσουμε να κάτσουμε ε, να τις κοιτάξουμε. Σημαντικό για μένα ήταν όσον αφορά τις συντάξεις, με πολλές εμπειρίες σε πολλά κράτη-μέλη, ε, που δεν είναι πολύ καλές, ε, ο κόσμος θα πρέπει να έχει συντάξει από τι οποίε μπορεί να ζήσει και γι' αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε τα κατάλληλα εργαλεία. Για να πάρουμε στα σοβαρά τους ηλικιωμένου, ε, θα πρέπει όχι απλά να μειώνουμε τα πάντα, αλλά να έχουν αρκετό εισόδημα ώστε να μπορούν να επιβιώσουν. Και αυτό θέλουμε να φαίνεται στην έκθεση αυτή δικαιοσύνη απέναντι στις διάφορες ε, γενιές. Δεν είναι να θεωρούμε ότι ο ο ηλικιωμένος κόσμος δεν μπορεί να εργαστεί. Σε πολλές επιχειρήσεις θεωρούνται ε, λόγω του μεγάλου κόστους ε, της εργασίας τους ε, σαν θεωρούνται μειονέκτημα. Αλλά αυτό είναι διάκριση λόγω ηλικίας. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι ακόμα ζωντανοί, μπορούν να εργαστούν, θέλουν να ε, εργαστούν και απαντούν συνεχώς αυτήν την διάκριση ότι δεν σας χρειαζόμαστε πια, πάει πέρασε. Και γι' αυτό λέμε, δημιουργήστε θέσεις απασχόλησης όπου οι νέοι και οι ηλικιωμένοι να μπορούν να εργαστούν μαζί. Να εποφεληθούμε από τη δημιουργικότητα των ανθρώπων αυτών. Αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεν θα πρέπει να λέμε ότι οι νέοι είναι υπερβολικά νέοι για να λάβουν κατάρτιση, ούτε θα πρέπει ε, να γίνονται διακρίσεις εις βάρος των ηλικιωμένων λόγων της ηλικία τους. Ε, υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι είναι εντάξει, ωραία, έχω κάποια προβλήματα υγείας, αλλά θέλω και μπορώ να εργαστώ. Ε, αυτά είναι παραδείγματα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Ε, δεν θα πρέπει λοιπόν να ε, θεσπίσουμε μια συγκεκριμένη ηλικία συνταξιοδότησης. Φρανσουάζ, αυτό ισχύει και όσον αφορά το νόμιμο όριο ηλικίας που αναφέρεις. Θα πρέπει να έχουμε τέτοιες ρυθμίσεις ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να μπορούν να συμφωνήσουν ε, για κάποιες ρυθμίσεις. Εγώ είμαι υπέρ ε, των κοινωνικών εταίρων, ε, υπέρ των συλλογικών συμβάσεων, αλλά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αλλά έχουμε εδώ πέρα ένα συγκεκριμένο τομέα. Όλο το ανέφερε. Το flexicurity είναι σημαντικό. Δεν θα πρέπει ξαφνικά να ξεχάσουμε την ασφάλεια και να έχουμε μόνο ευελιξία. Αυτό θα ήταν τελείω λάθο δρόμο. Συνάδελφε συμφωνώ. Όσον αφορά το εξάμεινο και το τετράμινο διαφωνούμε, αλλά με την ε, τροπολογία 228 Ε, αναφέρω ότι αυτό είναι σημαντικό στοιχείο. Η αμοιβαιότητα είναι σημαντική, θα πρέπει να βρούμε μια καλή ισορροφία. Και πιστεύω ότι αν χρησιμοποιήσουμε αυτή τη βάση, τότε θα προχωρήσουμε ε, καλά, Μέρι Χάρκιν, έχω συμφωνήσει με όλες τις τροπολογίες σας. Δεν υπάρχει ούτε ένα σημείο που θα ήθελα να αλλάξω. Και η τροπολογία 248 είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για την έκθεση αυτή. Ε, σας ευχαριστώ όλους. Θα προσπαθήσω να εκπονήσω συμβαστικές τροπολογίες. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου ε, που να θεωρούμε ότι μας βοηθάει να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Θα ψηφίσουμε για τις τροπολογίες που έχουν ολοκληρωθεί και ε, τις έχουμε διαπραγματευτεί. Στη δεύτερη μάλλον ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Καλές διακοπές λοιπόν και θα συνεδριάσουμε 13 Σεπτεμβρίου στις 3.